περάσουμε στην ε, ψηφοφορία στα πιο σοβαρά. Η πρώτη έκθεση αφορά την Ρωσία, την περίπτωση του ογιούμπ TTF. Οπότε έχουμε το ετοιμώντας 10 του αρχικού κειμένου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται υπέρ του ψηφίσματος στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην Αίγυπτο, εκτελέσεις στην Αίγυπτο. Εκτιμώντας G, μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία για το δεύτερο μέρος. Πέρας. Δεκτή. Εκτιμώντας M. Αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Υπέρ του ψηφίσματος, του σύνολό του, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην IT. Την παιδική δουλεία. Έχουμε ένα κοινό ψήφισμα, η τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το ψήφισμα στο σύνολό του υπέρ κατά αποχές δεκτό περνάμε τώρα στη σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής για την διαδικασία διοδότησης της ε, Ένωσης για τα ζυζανιοκτώνα. Την γνωρίζουμε αυτή τη σύνθεση. Δεν έχουμε λάβει κάποιες ε, τροπολογίες ε, επί της πρότασης αυτής της διάσκεψης των Προέδρων οπότε η πρόταση εγκρίνεται. Περνάμε στην επόμενη έκθεση. Θέλει κάποιος τον λόγο υπέρ της ε, απόφασης της Επιτροπής. Υπέρ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Φιέλνερ που ζήτησε τον λόγο για να εκφραστεί κατά της πρόταση αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα έλεγα πως υπάρχει πληθωρισμό εδώ πέρα ψηφοφοριών για να πάμε σε διαπραγματεύσεις με βάση μια εντολή η οποία ψηφίζεται στην Επιτροπή και όχι στην Ολομέλεια. Και αυτό είναι προβληματικό. Είναι λογικό εάν υπάρχει ευρεία συνένεση στην Επιτροπή επί της ουσίας, αλλά στην περίπτωση αυτή, στα σημαντικότερα θέματα αυτού του φακέλου, ε, η διαφορά ήταν τρεις ψήφοι. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούμε το ότι ψηφίζουμε σε μία επιτροπή χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις άλλες επιτροπές, όπως εδώ πέρα την ε, Επιτροπή Μεταφορών. Επί της ουσίας, βεβαίως, το θέμα αφορά λιγότερο το ποιες πληροφορίες θα πρέπει να δίνουν οι χρήστες φορτηγών για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, αλλά περισσότερο το πώς πληροφορίες θα δίνουν για να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι Κινέζοι ανταγωνιστές. Αλλά το πρόβλημα είναι άλλο. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να αποφασίσει την διαπραγματευτική έντολη του Κοινοβουλίου και όχι κατά κανόνα να το αποφασίζει αυτό η Επιτροπή Περιβάλλοντος ή οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή. πρέπει να καταψηφίσουμε αυτήν την εντολή χωρίς, ε, αφού δεν την έχουμε εξετάσει. Να σας ρωτήσω και πάλι. Υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι υπέρ της πρότασης της Επιτροπής. Θέλει κάποιος να μιλήσει υπέρ. Όχι. Μάλιστα. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της απόφασης κατά αποχές λοιπόν να το αρχή την ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται Λοιπόν, περνάμε στην επόμενη έκθεση, Dalton. Ο... Στίβενς, έχετε το λόγο για να μιλήσετε υπέρ της απόφασης. Thank you, President. Κυρία Χέλγα Στίβενς, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ο κύριος Ντόλτον κολλείεται και ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να παρουσιάσει ο ίδιο το θέμα αυτό. Ε, ο κανονισμό είναι σημαντικό βήμα για να κλείσουν κάποια παραθυράκια και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση τη εγκληματικότητα και να εξασφαλιστεί αποτελεσματική ανταλλαγή υπηρεσιών για προηγούμενε καταδίκε ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό για να εξασφαλιστεί εμπιστοσύνη και αμοιβαία αναγνώριση στα θέματα δικαστική συνεργασία. Και είναι σωστό να είναι ποιοτική η ανταλλαγή πληροφοριών για καταδίκες ε, ε, και υπηκόν τρίτο χώρο και υπηκόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με βάση το σημερινό σύστημα, η CIRS, εντοπίζουμε προηγούμενες καταδίκες για υπηκός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όχι για υπηκός τρίτων χωρών. Και χάρη στην έκθεση αυτή ε, διορθώνεται αυτό το, αυτή η έλλειψη. Και μάλιστα ή ε, πέρασε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ γιατί εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία μεταξύ των ε, δικαιωμάτων των ε, προσώπων αλλά και τη σωστή ενημέρωση για προηγούμενες καταδίκες. Επίσης, οι δικαστικές αρχές και οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να διεξαγάγουν το έργο τους με τα κατάλληλα εχέγγυα ότι τα στοιχεία για τι καταδίκες αυτέ που έχουν γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσιτά μόνο υπό συγκεκριμένου όρου. Επίση, προβλέπονται απαραίτητε εγγυήσει για την πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία. Και αυτό ακριβώ πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίζονται τα συγκεκριμένα εχέγγυα ό,τι αφορά την πρόσβαση τέτοιων πληροφοριών για προηγούμενε καταδίκε. Καταδικαστικέ αποφάσει. Ο κύριο Πιμέντα Λόπε είναι κατά. Ναι, το είπα και στο Προεδρείο και το θέσαμε στην Ολομέλεια. Έχουμε μια έκθεση που υπευλήθη μόνο στα αγγλικά, χωρίς καμία μετάφραση, κάτι που συνιστά κατάφορη, παραβίαση της αρχής της πολυγλωσσίας. Ε, και αυτό οφείλεται εν μέρη λόγω και της συρρήκνωσης του προπολογισμού, της περικοπής των εξόδων και για τις μεταφράσεις. Ε, με αποτέλεσμα να έχουμε την απαράδεκτη κατάσταση, το έγγραφο της έκθεσης να υποβάλλεται μόνο σε μία γλώσσα, στα αγγλικά. Όπως ε, μου υπενθυμίσει η Γραμματεία, τώρα αποφασίζουμε για την απόφαση της Επιτροπής και όχι για το κείμενο της έκθεσης δόλτον Με ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην έκθεση Γκαρδιασάμπαλ Ρουβιάλ με θέμα το Ταμείο Εγγύσεων για τις Εξωτερικές Δράσεις. Ονομαστική ψηφοφορία για την τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενη έκθεση Γουαρδία Σάβολα Ρουμπιάλ για την εγγύηση Ευρωπαϊκής Ένωση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τροπολογία 64 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρίτη έκθεση Γκαρδία Σάπαλ Ρουμπιάλ για την ετήσια έκθεση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τροπολογία 6 με ονομαστική κλίση, άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορία. Απορρίπτεται η τροπολογία 6. Τροπολογία 7. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται και η 7. Τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. και το σύνολο του ψηφίσματος με ονομαστική κλίση άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην παρούσα κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 2 άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Άρχεται ψηφοφορία. ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Για την παράγραφο 8 έχουμε μια προφορική τροπολογία. Περιλαμβάνεται στον κατάλογο ψηφοφορίας. Αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να ζητήσω από την συντάκτρια την κυρία Κουμπούλα Νάτρη να την παρουσιάσει. Αγαπητοί συνάδελφοι, αφορά την παράγραφο 8 που αφορά την πολιτική πίεση στους ε, δημοσιογράφους. Προτείνω να προτείνουμε καλή την Τουρκία να ε, αποσύρει τις κατηγορίες κατά του, της Άιλα Αλμπαράκ, φιλαδό τουρκικής κα, ε, καταγωγής, που καταδικάστηκε ερήμην. Μάλιστα, ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η προφορική τροπολογία. Παράγραφος 10 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Παράγραφος 13 σε δύο τμήματα. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη μη αρχικό κείμενο υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το σύνολο του ψηφίσματος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στο επόμενο ψήφισμα που αφορά την κατάσταση στη Βενεζουέλα. Έχουμε ένα κοινό σχέδιο ψηφίσματος, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Επόμενο θέμα, κατάσταση υπηρεσίας αρρωγής και έργων των Εθνών υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τελευταίο θέμα, ε, διατάξει τη θερινή ώρα, τροπολογία 1, ποιος είναι υπέρ, έκθεση που θα επηρεάσει την καθημερινότητά μας κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 4 Άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 2 υπέρ μάλλον άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 2 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και το σύνολο του ψηφίσματος υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες.